Γιώργο. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Πρόεδρε των Επιτροπών, αξιότιμοι συνάδελφοι από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με μεγάλη χαρά και τιμή εμφανίζομαι ενώπιόν σας. Γνωρίζω το χαρτοφυλάκιο το οποίο θα επομιστώ εάν εγκριθώ ως Επίτροπος. Έχει σημαντικό αντίκτυπο για την καθημερινή ζωή όλων των ατόμων που βρίσκονται σε αυτή την αίθουσα και των 500 εκατομμύριων πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό με μεγάλο ενθουσιασμό αλλά και με ισχυρό αίσθημα ευθύνης που ζητώ την έγκρισή σας για να είμαι η Επίτροπος Δικαιοσύνης, Καταναλωτών και Ισότητας των Φίλων. με ενθουσιασμό πιστεύω όλοι μαζί μπορούμε πραγματικά να κάνουμε τη διαφορά. Όπως όλοι, όπως όλοι από εσά είμαι στην πολιτική γιατί θέλω να κάνω μια συμβολή στην κοινωνία. Θέλω να αφήσω τη σφαγίδα μου στις προσπάθειες να βελτιωθεί η ζωή των ανθρώπων και να το επιτύχω μέσα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένας πιο γνωστός τσέχος πολιτικός, πιο γνωστός από μένα, βρέθηκε το 2000 ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και είπε το εξή. Οι κέρυες ευρωπαϊκές αξίες έχουν διαμορφωθεί από την ιστορία, την πνευματική ιστορία της Ευρώπης και έχουν μεγάλη σημασία για όλο τον κόσμο. Είναι ο σεβασμός για το άτομο και τις ατομικές ελευθερίες. Το, τα δικαιώματα του ατόμου και την αξιοπρέπειά του. Αξιοπρέπειά του. Η αρχή της αλληλεγγύης, η ισότητα ενώπιον του νόμου, το κράτος δικαίου, η προστασία των εθνοτικών μειονοτήτων, οι δημοκρατικοί θεσμοί, ο διαχωρισμός των εξουσιών, ο πολιτικός πλουραλισμός, ο σεβασμός για την ιδιωτική περιουσία και την ελευθερία του επιχειρήν, μια οικονομία, ε, μια ε, οικονομία της αγοράς και κοινωνία των πολιτών. Ο Βάτσλαβ Χάβελ ήταν πολύ μπροστά από την εποχή του όταν έκανε αυτή την ομιλία. Η δική μου λοιπόν δέσμευση ενώπιόν σας είναι να προσπαθήσω να πραγματώσω αυτές τις βασικές ευρωπαϊκές αξίες και αρχές που τόσο καλά παρουσίασε ο Βάτσλαβ Χάβελ και να εξασφαλίσω ότι θα τύχουν σεβασμού. Γιατί αυτές είναι οι αρχές τις οποίες και εγώ έχω ενστερνιστεί. Το χαρτοφυλάκιο της δικαιοσύνη των καταναλωτών και της ισότητας των φύλων θα πρέπει να βοηθήσει να, να υλοποιηθούν αυτές οι αρχές με το να δημιουργήσει γέφυρες μεταξύ των ευρωπαϊκών νομικών συστημάτων. Θα πρέπει να ενισχύσει την οικονομική ανάπτυξη γιατί μια ορθή, υγιής και αξιόπιστη δικαιοσύνη είναι προϋπόθεση για ένα καλό επιχειρηματικό πλαίσιο όπου μπορεί να λειτουργήσει το διαμεθοριακό εμπόριο. Πάνω απ' όλα το χαρτοφυλάκιο αυτό έχει να κάνει με τη δημιουργία μιας ε, κοινωνίας όπου τα άτομα βρισκόνται στο κέντρο. Μέσα σε όλες τις δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να δώσουμε επιλογές στους ανθρώπους, να προστατεύσουμε τα δικαιώματά τους και να αυξήσουμε την εμπιστοσύνη τους. Αν αφήσουμε κατά μέρος την πολυπλοκότητα και τις νομικές έννοιες, όλες οι προτάσεις που θα γίνουν από την Κομισιόν που έχουν γίνει από την Κομισιόν και θα γίνουν από την Κομισιόν για τα θέματα αυτά επιζητούν αυτά τα τρία στοιχεία. Περισσότερες επιλογές, περισσότερη προστασία και περισσότερη εμπιστοσύνη. Στο έργο αυτό θα προσπαθήσω να λάβω υπόψη τα συμφέροντα όλων των πολιτών μας. Είναι μια ευκαιρία να μπορέσουμε να συνενώσουμε όλα αυτά τα στοιχεία του χαρτοφυλακίου μαζί. Τα επόμενα πέντε χρόνια, αγαπητά μέλη του Κοινοβουλίου, θέλω να κάνω τη διαφορά στους τρεις αυτούς τομείς που προανέφερα. Καταρχήν με το να εξασφαλίσω ότι υπάρχει περισσότερη επιλογή για τα άτομα. Σε πρακτικούς όρους, τι σημαίνει αυτό σημαίνει ότι θα έχουν το δικαίωμα να αποφασίσουν που θέλουν να ζουν και να εργάζονται και να έχουν πλήρη σεβασμό για την ελευθερία διακίνησής του. Πρέπει πράγματι να αντιμετωπίσουμε τις καταχρήσεις όπου υπάρχουν, αλλά το θεμελιώδες δικαίωμα για την ελεύθερη κυκλοφορία δεν θα πρέπει να τεθεί ένα αμφιβόλο. Επίσης, θα πρέπει οι πολίτες μας να ζουν εκεί που θέλουν να ζουν, χωρίς διακρίσεις με ασφάλεια, χωρίς φόβο παρενοχλήσεων και βιαίων επιβολών. Ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τη δυνατότητα να βελτιώσει τα δικαιώματα αυτά, ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα πρέπει να παραμελήσει να το κάνει αυτό. Αυτό σημαίνει να σπάσουμε το, τη γυάλινη οροφή ώστε οι γυναίκες μπορούν να ανέλθουν σε θέσεις ε, ευθύνης με την ίδια δυνατότητα όπως και οι άνδρες και να έχουν ίση αμοιβή για ίση εργασία. Θα υπερασπιστώ λοιπόν τις προτάσεις που έχουν να κάνουν με τα δικαιώματα των γυναικών. Αυτό επίσης σημαίνει ότι θα πρέπει και οι καταναλωτές να έχουν τη δυνατότητα να επιλέγουν όντας πληροφορημένοι και επίσης να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίε που τους δίνει η ψηφιακή επανάσταση και να μπορούν να ενσωματώσουν τις επιλογές τους και σε αυτή τη ψηφιακή οικονομία. Επίσης, να έχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν μια ε, σχέση συμβίωσης, να παντρευτούν και να υπάρχει μια οικουμενική αναγνώριση των, αντίστοιχων νομικών αποφάσεων και των δικαιωμάτων ιδιοκτησία που εκπηγάζουν από αυτές. Πρέπει λοιπόν να προστατεύσουμε και τα δικαιώματα των πολιτών μας. Θα βοηθήσω τον Αντιπρόεδρο κύριο Τίμερμαντς και να του δώσω την πλήρω υποστήριξή μου για τη διατήρηση του κράτους δικαίου και την, ε, το σεβασμό της χάρτας θεμελιωδών δικαιωμάτων, ώστε να εξασφαλίσουμε ότι οι απαραίτητοι διασταυρούμενοι έλεγχοι οι οποίοι ισχύουν στις δημοκρατίες μας θα πρέπει να διεχάρουν πλήρους σεβασμού και εφαρμογής και να εξασφαλίσω επίσης ότι η πρόσβαση της Ευρωπαϊκής, προσχώρηση συγγνώμη, της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ε, Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης θα πραγματοποιηθεί το ταχύτερο δυνατό. Θέλω επίσης να εξασφαλίσω ότι θα τύχουν προστασία στα δικαιώματα των πολιτών μέσα από την ταχεία έγκριση μιας μεταρρύθμισης για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και ότι οι Ευρωπαίοι θα την χάνουν ίσης προστασίας και στις Ηνωμένε Πολιτείες. Θέλω να εξασφαλίσω επίση ότι οι εθνοτικές μειονότητες όπως η Ρωμά θα προστατεύονται από τον αποκλεισμό και τις διακρίσεις και θα ενσωματωθούν περαιτέρω στην κοινωνία μας. Θέλω επίση να προστατεύσω τα πιο ευάλωτα μέλη της κοινωνίας μας αυτό σημαίνει να διατηρήσουμε τα δικαιώματα του παιδιού, ιδίως στο διαδίκτυο, και να εξασφαλίσουμε ότι τα παιδιά έχουν το δικαίωμα σε δίκαιες δίκης όταν είναι ε, υπο, υποψία, όταν είναι ύποπτη σε ποινικέ διαδικασίες. Θέλω να υπάρξει ένα αποτελεσματικό γραφείο εισαγγελέω στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να προστατεύσει την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον προπολογισμό της από απάτες. Θέλω να υπάρξει βιώσιμη και ε, στεναρή ε, αντιμετώπιση των εξωστομέων. Εταιρική ευθύνη που έχει να κάνει με τη σωστή παρουσίαση πληροφοριών στους καταναλωτές και την προστασία τους. Θα εργαστώ με την Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή για να εξασφαλίσω ότι και οι κανόνες για τα μπόνους των, ε, των τραπεζικών στελεχών εφαρμόζονται πλήρως. Η προστασία των καταναλωτών σημαίνει επίση ότι θα πρέπει να είναι ασφαλή τα προϊόντα που χρησιμοποιούμε. Θέλω να υπάρξει ταχεία εφαρμογή, έγκριση και εφαρμογή του πακέτου για την εποπτεία της αγοράς και την προστασία των καταναλωτών. Τέλος, όταν μιλάω για προστασία, σκέφτομαι την κατάσταση των γυναικών που είναι θύματα βία μέσα στην οικογένεια και τις ε, απάνθρωπες πρακτικές ε, γυναικείου σεξουαλικού ακροτηριασμού. Όλα αυτά είναι απόλυτα ασύμβατα με τις αξίες και τις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα βήματα τέτοιας βίας χρειάζονται να έχουν την υποστήριξή μας. Θέλω να δημιουργήσω και εμπιστοσύνη μεταξύ των νομικών συστημάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να είμαστε ενωμένοι στην πολυμορφία μας, αλλά θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι οι διαφορετικές μας ιστορικές και πολιτιστικές παραδόσεις δεν είναι εμπόδιο στην ελευθερία, τη δικαιοσύνη ή την εσωτερική αγορά. Οι πολίτες της Ευρώπης χρειάζονται να έχουν εμπιστοσύνη στο νομικό σύστημα της, Ευρω... της χώρας τους και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτά τα συστήματα θα πρέπει να εμπνέουν εμπιστοσύνη. Η αμοιβαία αναγνώριση, όπως στην περίπτωση του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Συλλήψης, συλλήψεως ή η εφαρμογή νομικών αποφάσεων από άλλα κράτη-μέλη μπορούν να λειτουργήσουν μονάχα επί τη βάση της απαραίτητης εμπιστοσύνης. Όταν αυτό είναι απαραίτητο θα χρειαστούμε περαιτέρω συντονισμό, θα χρειαστούμε ελάχιστα πρότυπα που να ισχύουν σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, τόσο στις αστικές όσο και στις ποινικέ υποθέσεις. Χρειαζόμαστε επιπλέον να βελτιώσουμε και την αμοιβαία γνώση των νομικών συστημάτων ημέν των δε. Μπορούμε λοιπόν να έχουμε και μια νέα όθηση για την εκπαίδευση των νομομαθών που είναι απαραίτητη για να μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν τα εργαλεία που θέλουμε να θέσουμε σε εφαρμογή και να επιτύχουν επίσης το στόχο του αυτά τα μέτρα. Πιστεύω στην ηλεκτρονική ε, δικαιοσύνη που μπορεί να επιταχύνει την αποδότηση τη δικαιοσύνη και να βελτιώσει την πρόσβαση των πολιτών και των επιχειρήσεων στη δικαιοσύνη. Είναι ο στόχο μου να αναβαθμίσω το εργαλείο αυτό σε ένα πιο διαδραστικό εργαλείο για όλου. Θέλω επίση να εξασφαλίσω ότι οι καταναλωτέ θα έχουν εμπιστοσύνη στι αγοραπολισίε στι οποίε επεμβαίνουν, γνωρίζοντα ότι θα έχουν και δυνατότητα νομική θεραπεία όταν το πράττουν σε μια άλλη χώρα εκτό από τη δική του. Και επίση θέλω να προωθήσω τη δυνατότητα να υπάρχουν πιο εύκολα πρόσφυγες για τα θέματα αυτά και να προωθήσω την εναλλακτική επίλυση διαφορών. Θα ήθελα επίσης να υπάρξει και, εάν είναι απαραίτητο, συλλογική θεραπεία σε περιπτώσει που χωρεί κάτι τέτοιο. Επίσης πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση στις εκτελεστικές εξουσίες, ώστε να μην πέφτουν θύματα οι πολίτες μας. Σε συγκεκριμένους τομείς θα πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ κρατών μελών ώστε να υπερασπιστούμε τα δικαιώματα των καταναλωτών. Έντιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Να προσθέσω και μια προσωπική νότα τώρα. Πριν από 8 χρόνια, πριν από 8 χρόνια ήμουν φυλακισμένη στην τσεχική ε, δημοκρατία γιατί ήμουν θύμα μιας άδικης δικαστικής διαδικασίας. Αυτό ήταν κάτι που με σοκάρισε. Εγώ δεν πίστευα ποτέ ότι θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο, να φυλακιστεί κάποιο χωρί να υπάρχουν στοιχεία πραγματικά σε βάρος του. Και μετά από κάποια χρόνια αποδείχθηκε ότι ήταν χαλκευμένη η κατηγορία εναντίον μου και ήταν απόλυτα παράνομη. Αυτός ήταν ο τρόπος με τον οποίο εγώ βλέπω τώρα τη δικαιοσύνη. Μετά από αυτό το σοκ θα ήθελα να εξασφαλίσω ότι η δικαιοσύνη μπορεί πράγματι να λειτουργήσει και γι' αυτό το λόγο αυτό άρχισα να εργάζομαι ε, ως νομομαθής. Έγινα φοιτήτρια νομικών στην Πράγα και το έπραξα αυτό με στόχο να γίνω νομομαθής και να έχω μια νέα αποστολή γιατί και η εργασία που είχα στο παρελθόν ήταν σε ένα χώρο που το όνομά μου είχε σπηλωθεί. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο τώρα μετά από τόσα χρόνια με έχει σημαδέψει αυτή η εμπειρία και όταν έρχομαι αντιμέτωποι με αδικίες νιώθω την ίδια αγανάκτηση. Γι' αυτό θέλω να υπάρξει μια κοινωνία όπου οι πολίτες μας έχουν προστασία, επιλογή και εμπιστοσύνη. Δεν πρέπει να χάσουμε την εμπιστοσύνη μας ότι στο τέλος θα επικρατήσει η δικαιοσύνη. Τουλάχιστον στη δική μου περίπτωση έγινε αυτό πραγματικά. Και το νομικό σύστημα της Τσεχίας μου έδωσε μια αποζημίωση και το όνομά μου έχει ε, καθαριστεί από τις κατηγορίες αυτές. Αγαπητοί συνάδελφοι, χαίρομαι πάρα πολύ που μπορεί να κληρονομήσω ένα όγκο έργου που ήταν πάρα πολύ σημαντικός και που μου έχει κλειδωτηθεί από τους προκατόχους μου, όπως η Βιβιάνε Ρέντινγκ, που έθεσε μία σειρά από προτάσεις για τα ζητήματα αυτά. Έρχομαι από τον κόσμο της περιφερειακής πολιτικής, των διαρθωτικών ε, ταμείων, των σχεδίων, των χρονοδιαγραμμάτων κτλ. Ως Υπουργός Περιφερειακής Ανάπτυξης ε, είναι η τελευταία μέρα που είμαι υπουργό γιατί αύριο θα παρετηθώ. πιστεύω ότι μπόρεσα να εφαρμόσω μια συγκεκριμένη στρατηγική στην ψυχή δημοκρατία που θα καλύψει την επόμενη δεκαετία. Εγώ συμμερίζομαι απόλυτα και θα υποστηρίξω τη νέα προσέγγιση που υποστηρίζει ο πρόεδρος Γιούγκερ και οι πολιτικοί του υποστηρικτές γιατί πιστεύω ότι αυτή είναι ακριβώς η προσέγγιση που θέλω να πάρω στο νέο μου αυτό ρόλο. Πρέπει να ξεπεράσουμε τα στεγανά να έχουμε συνεργασία των επιτρόπων πέρα από στενά χαρτοφυλάκια επί τη βάση των αρχών που ανέφερα προηγουμένω. Είμαι εκλεγμένη βουλευτής από το, στο Τσεχικό Κοινοβούλιο για τις τελευταίες μου μέρες. Είμαι πολιτικός από την κοινωνία των πολιτών και θέλω να ενισχύσω αυτό το χώρο. Αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Δεν μπορώ να αναφέρω όλα τα θέματα τα οποία θα τύχουν της προσοχής μου σε αυτό το τόσο συναρπαστικό χαρτοφυλάκιο αλλά έχουμε κοινού στόχους και πιστεύω ότι μπορούμε από κοινού να επιτύχουμε αυτούς τους στόχους. Ας ξεκινήσουμε με το να έχουμε θετικά αποτελέσματα που περιμένουν οι Ευρωπαίοι πολίτες από μας για την μεταρρύθμιση των κανόνων για την προστασία δεδομένων, για τον ε, Ευρωπαϊκό ε, Εισαγγελέα, για την οδηγία για τα προϊόντα, για την οδηγία Women on Board, Θέλω λοιπόν μαζί σας να αναπτύξω μια νέα ατζέντα για τα επόμενα χρόνια που να συνδέουν όλα τα στοιχεία του χαρτοφυλακίου μου. Αν το πετύχουμε αυτό, θα μπορέσουμε να έχουμε μια εσωτερική αγορά που να είναι θετική και για τις επιχειρήσεις και για τους καταναλωτές. Να επαναλάβω και πάλι. Θέλω να υπάρχει περισσότερη επιλογή, περισσότερη προστασία και μεγαλύτερη εμπιστοσύνη. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.